So um, Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτελικών Ελευθεριών και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών υπό το άρθρο 55. Να καλώς ορίσω τα μέλη της Επιτροπής ΦΑΜ και την Πρόεδρο ασφαλώς της Επιτροπής. Αν θα θέλετε να κάνετε μία σύντομη εισαγωγή, παρακαλώ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν στις 4 Μαρτίου να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, συνθήκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και εγκρίθηκε το βήμα αυτό. Έγινε και μία δήλωση και μία ένα σχέδιο έκθεση. κατατέθηκαν 380 τροπολογίε στην έκθεση και με χαρά θα δώσω τώρα το λόγο στην Βίλια, την Πρόεδρο τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μωράε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνθήκη τη ε, Κωνσταντινούπολης. Μεγάλο βήμα για την ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και Έχουμε διοργανώσει δύο ακροάσεις, δημόσιες ακροάσεις, ακούσαμε και παρουσιάσεις του, της ενδιάμεσης έκθεσης και όπως είπατε πλέον έχει έλθει η στιγμή εξετάσεις των τροπολογιών για το σχέδιο. Να δώσω το λόγο στη συνσυγητρία, την κυρία Μπονιφέη. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε έχω, θα ήθελα να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω τον Σκιώδη και όλους τους, άλλες, όλους τους άλλους που κατέθεσαν τροπολογίες. Και εμεί είμαστε περιορισμένοι σε ό,τι αφορά τις 6.000 χαρακτήρες που ήταν το όριο για την το πρώτο σχέδιο. Και εγώ κατέθεσα ε, τροπολογίε και προσωπικά και από πλευράς της ομάδας μου να ευχαριστήσω και όσους με υποστηρίξαν, να ευχαριστήσω και την κυρία Κορατσαμπέλτ ε, που μαζί επίσης ε, καταθέσαμε τροπολογία. Οι πιο πολλές μας βρίσκουν σύμφωνοι και ε, κινείται προς τη σωστή κατάσταση για να υπάρξει συνένεση σε κάποια βασικά θέματα προκειμένου να ξεπλουγκάρουν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα αίτια και τις συνέπειες της ανισότητας των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν καθολικές λύσεις σε αυτά τα καθολικά προβλήματα. Και επίσης να αλλάξει και η νοοτροπία σε όλη την ε, κοινωνία μέσω της παιδείας, της σεξουαλικής εκπαίδευσης και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πρόκειται για μια καταπολέμηση όλων των στερεοτύπων ε, μέσω των κοινωνικών μέσων, του τύπου και το καθεξής. Επίσης, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, στην προστασία και στην παρακολούθηση και συμφωνώ μαζί σα ότι αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα θα πρέπει να τιμωρούνται και οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν όλη την υποστήριξη του δικαστικού συστήματο. συστήματος. Επίσης, ε, θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, εκ νέου θυματοποίηση των θυμάτων και επίσης ε, να υπάρχουν και ανθρώπινοι αλλά και οικονομικοί πόροι για να εφαρμοστεί η συνθήκη. Γιατί το διακύβευμα είναι μεγάλο. Θα θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε όσοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νομοθετική πράξη. Φαίνεται βασικό αυτό το βήμα και θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα νομοθέτημα, ίσως μια οδηγία, η οποία θα μας βοηθήσει να συμφωνήσουμε επί κοινών όρων για τα εγκλήματα κατά των γυναίκων και να επιτρέψει την εφαρμογή της συνθήκης και χαίρομαι που και άλλοι συναδελφοί με υποστηρίζουν και επίσης ε, να σας υπογραμμίσω τις τροπολογίες που ζητούν τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συντονιστή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και υπάρχουν ανεξάρτητα όργα, θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα όργα τα οποία θα δημιουργηθούν από τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και η Γκουέ και η Άλδε και οι σοσιαλδημοκράτες μας υποστηρίζουν και είμαι βέβαιη θα μας υποστηρίξουν και άλλες ομάδες ένα άλλο θέμα το θέμα της παραγράφους κατά, για την ε, πολλαπλή διακριτική μεταχείριση γυναίκες ε, μετανάστες, ανάπηρες, ρομ, λεσβίες όλα αυτά λοιπόν ε, θα πρέπει να λεφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά και τη διάσταση της ομοφοβίας, ό,τι αφορά τη διάσταση του ρατσισμού και τέλος να υποθυμίσουμε τις τα προβλήματα των γυναίκων, των γυναικών με αναπηρία. Οι πιο πολλοί από εσά το υποστηρίζουν και η τροπολογία περιθμού 40 τη συνσηγήτριας αναφέρεται στην ε, διάσκεψη των ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Να σα υπενθυμίσουμε ότι οι γυναίκε αυτέ με αναπηρία θα πρέπει να προστατευτούν από τη βία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη. Η κυρία Στίβεν. Ε, ανέφερε ότι όλα τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διάκριση, είτε πρόκειται για εθνοτικό, θρησκευτικό, σεξουαλικό υποβάθρο. Επίσης, να σας αναφέρω την τροπολογία μου για την έκτρωση και την τροπολογία της κυρίας Κούνεβα και της κυρίας Μπόργκ επίσης για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει να αναφέρετε σε κάποιες περιπτώσεις όταν πρόκειται για βιασμούς ε, και εγκυμοσύνες που προκύπτουν πρόκειται για ένα έγκλημα βίας κατά των γυναικών. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νόμιμες εκτρώσεις οι γυναίκες, σε νόμιμες αμπλώσεις. Αυτό θα είναι πέραν από κάθε συζήτηση. Γιατί θεωρείται βία και η άρνηση της άμβλωσης. Θα πρέπει να σας αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα και δεν βλέπω κανένα άλλο τρόπο να ακολουθήσουμε το θέμα αυτό. Ιδιαίτερα σήμερα, όπου βλέπουμε μέτρα αντίδραση από όλη την Ευρώπη. Να μην σα επενθυμίσω καν τι γίνεται στην Πολωνία. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην ουσία του θέματο ότι αν δεν προασπίσουμε το δικαίωμα στην άμβλωση, ποιο θα το πράξει. Να μην ξεχνάμε και τις γυναίκες που διαδίωσαν στην Πολωνία κατά τη κυβέρνηση Και τέλο υπάρχουν και άλλε τροπολογίε οι οποίε παρουσιάζουν προβλήματα και τι οποίε δεν θα υποστηρίξω αυτή για παράδειγμα που λυπούνται και για την προσχώρηση στη συνθήκη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούν ότι είναι ίσονος σημασία και ότι αποτελεί ένα θέμα μόνο που θα ε, βοηθήσει μόνο τους μετανάστες αναφέρονται στι γυναίκε μόνο μητέρα, για παράδειγμα. Μαζί με τη σκιώδη εισηγήτρια συναντηθήκαμε στι 18 Μαου, συνεργαστήκαμε επικοδομητικά, συμφωνήσαμε επί τροπολογιών και σε ό,τι αφορά τι ανάπηρε γυναίκε και πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτέ τι γυναίκε να αμυνθούν κατά τη βία και το θέμα τη πολλαπλή ε, θυματοποίηση το αναφέραμε. Σε ό,τι αφορά επίση ε, τι συνέπειε σε ψυχολογικό, οικονομικό, σεξουαλικό, πνευματικό επίπεδο. Επίσης, ε, τα παιδιά τα οποία είναι θύματα οικογενειακή βίας, ε, αναφερθήκαμε στην κατάσταση στην κοινωνία και το πώ θα πρέπει να γνωριστεί η, τα δικαιώματα των γυναικών σε πλήρες επίπεδο και τέλο ότι οι γυναίκες δεν ε, προστατεύονται επαρκώς σε όλη την Ευρώπη λόγω της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης και Μία, τονίσαμε επίσης την έλλειψη νομοθετικής ε, πρόβλεψης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σωστή πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα και συμφωνήσαμε και για τα μέτρα αυτοάμυνας, για να αποφευθεί η θυματοποίηση των γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση βέβαια να μην αναγνωρίζεται αυτό ως δικαιολογία για πράξεις βίας και να σας πω επίσης ότι λάβουμε υπόψη και μία νέα μορφή βίας στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο. Ε, η ειδωνοβλεψία. Και ε, αναζητούμε λοιπόν μια συμφωνία για τις σχετικές ε, ρυθμίσεις και σε ό,τι αφορά άσυλο και μετανάστευση να σας πω ότι ως μέλος της Επιτροπής ΛΥΠΕ είμαι προφανώς ε, πολύ ευαίσθητη σε τέτοια ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, να ψηφίσουμε 10-11 Ιουλίου την έκθεση αυτή στη ΛΥΠΕ και στη ΦΑΜ και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με την εισηγήτρια και είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρουμε να λυθούμε στο ύψο για να μην απογοητεύσουμε τι γυναίκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει με θετικό και επικοδομητικό τρόπο να επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα με αυτά που διατείνονται όλα τα λαϊκιστικά κινήματα. Και τέλος, να κλείσω εν συντομία με τη συμφωνία που δημιουργήθηκε, που προέκυψε από τις 11 Μαΐου του 2017 και βάσει της οποίας ε, προσχώρησε η Ένωση στην ε, Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρόκειται για αρμοδιότητα το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργασία δικαστική για θέματα ποινικά και ε, συμφωνία για την ε, ε επιστροφή των ε, μεταναστών. Αναρωτιόμαστε και θα το τονίσουμε αυτό στην έκθεση για τις νομικές συνέπειες και θα πρέπει να κατανοήσουμε τις συνέπειες και τα αίτια τις εφαρμογή της συνθήκης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς θα σας τηρήσουμε ενήμερους με μια σχετική γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, λέγει Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Πέντε λεπτά έχετε στη διάκριση σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφο Κριστίνη, η συγγήτρια στη ΛΥΜΠΕ. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Για μένα ε, αυτή η συμφωνία, ε, μάλλον ε, η σύμβαση μάλλον του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι αυτή που είναι η σπονδυλική στήλη για την περάσπιση των γυναικών. Θέλουμε να δώσουμε φωνή στις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα βίας στην Ευρώπη και ε, να πούμε ότι η ενδοκιογενειακή βία είναι σοβαρό έγκλημα και πρέπει ως τέτοιο να τιμωρείται. Μιλάμε για την βία των ανδρών κατά των γυναικών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί όχι επειδή είσαι σύζυγος, όχι επειδή με εγκατέλειψε ή επειδή είσαι ντυμένη με κάποιο τρόπο ή επειδή πίνεις αλκοόλ ή επειδή ζηλεύεις. Δεν υπάρχει καμία θρησκεία παράδοση ή πολιτισμός που να μπορεί να δικαιολογεί το ξύλο, το δολοφονία, το βιασμό και ένα σωρό άλλα εγκλήματα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι να, το σημαντικό να ζητήσουμε από όλα τα κατεμέλη να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση και να την εφαρμόσουν πλήρως. Επίσης, όπως σωστά είπε η Κριστίν, να ε, πάμε πιο μακριά από την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο. Είμαστε ευγνώμονες στην Προεδρία της Μάλτας που πέτυχε αυτό το πρώτο τουλάχιστον να υπογράψουν ε, για την πρόσβαση της Ένωσης στην ε, Σύμβαση, αλλά λυπούμεθα που έχει περιορίσει τις αρμοδιότητες θα πρέπει να πιέσουμε ώστε να αυξηθούν με την επόμενη μας ε, Προεδρία. Αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το σεξισμό, τα στερεότυπα, το στιγματισμό, το, το στίγμα, να αλλάξει γενικά η νοοτροπία απέναντι στις γυναίκες και να συνεχίσουμε να προωθούμε την ισότητα των φύλων, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος μακροπρόθεσμα να έχουμε αποτέλεσμα για την, στην εκρίζωση της βίας κατά των γυναικών. Τώρα, για τις τροπολογίες, που είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, έχουμε 318 τροπολογίες. Η Κριστίν ήδη είπε πολλά οπότε εγώ θα είμαι σύντομη. Έχουμε συμπεριλάβει μετά από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων όλες τις προτάσεις ε, που προήλθαν από τους ε, συνάδελφους για τις ανάπηρες γυναίκες, για τις κατευθύντες γραμμές προς τα κατημέλη, ώστε να τους βοηθήσουμε να εφαρμόσουν τη σύμβαση της ε, Κιωσταντινούπολης, να την κυρώσουν και επίσης γίνεται και ειδική αναφορά στην ευάλωτη χαρακτήρα των παιδιών καθώς και τη νέα βία, την επιγραμμική μέσω δικτύων δηλαδή. Ε, ως εισηγήτρια γυναίκα και ως ομάδα του ΕΛΚ θα ήθελα να ζητήσω από όλους να, να, να είστε προσιλωμένοι στο θέμα της βίας κατά των γυναικών και στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης γιατί το κείμενο πρέπει να είναι οξύ ε, και ε, επί του θέματος και κέριο για να έχει αντίκτυπο. Να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να να τα πείσουμε βασικά ότι πρέπει να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο νομικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τη βία, να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία και να προστατεύσουμε τα θύματα. Με την Χριστίνα επίσης συμφωνήσαμε για τη δημιουργία ενός νομικού μέσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ω επόμενο βήμα αφού θα έχουμε πετύχει αυτό το κομμάτι της σύμβαση ε, τη Κωνσταντινούπολη, ώστε να έχουμε όλα τα δυνατά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα επίση σε αυτή την έκθεση να μην πούμε θέματα, ε, να μην μιλήσουμε για θέματα που είναι εκτό ή να στηρίξουμε τροπολογίε που κινδυνεύουν να διχάσουν ε, την εξαιρετική συνένεση που έχουμε. Αναφέρεται το θέμα της άμβλωσης. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η απόψή μου εδώ. Είμαι υπέρ της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση και να ρωτήσουμε και τους εμπειρογνώμονε ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση αναφέρει το θέμα της καταναγκαστικής άμβλωσης ω μορφή βία. Δηλαδή, αν σε αναγκάσει κάποιος να κάνει έκτρωση, αυτό είναι βία κατά της γυναίκας. Κάθε μορφή άμβλωσης δεν περιλαμβάνεται, οι υπόλοιπε μάλλον ε, μορφές άμβλωσης δεν περιλαμβάνονται εκεί και μάλιστα δεν είναι δική μας αυτή η σύμβαση και εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα του αν ε, είμαστε υπέρ ή όχι της άρνησης της άμβλωσης. Ε, το θέμα είναι να ακολουθήσουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τροπολογίες των συναδέλφων να εστιάζονται στην άρνηση. Παρακαλώ όμως μην το με παρεξηγήσετε και μην το χρησιμοποιήσετε για να διασπάσετε τη συνένεση. Μιλάμε για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Για αυτή την ε, σύμβαση μιλάει η έκθεση. Δεν ανοίγουμε συζήτηση για την άμβλωση. Έχουμε ένα σωρό άλλα φόρα όπου μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και είναι θέμα το τι κάνει το κάθε κράτος, τι κάνει ε, ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την θέση. Δεν θα στηρίξω τις τροπολογίες λοιπόν που είναι εκτός θέματος. Πολλές ε, δε τροπολογίες έχουν κατατεθεί από το ίδιο το ΕΛΚ και δεν θα τις υποστηρίξω ως εισηγήτρια του ΕΛΚ. Με τους σκιώδεις έχουμε συμφωνήσει σε διάφορες πολύ καλές συμβιβαστικές ε, έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τη συνεργασία για την εξέβρεση και άλλων συμβιβαστικών και να πω σύντομα τι έχουμε περιλάβει. Αν, ε, γυναίκες με ειδικέ ανάγκες, ευάλωτες ομάδες είναι αντικείμενα πολλαπλών διακρίσεων, σημασία καταπολέμησης ατιμορρησίας και δίκης ε, των δραστών, σημαντικός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, στην διεύθυνση των καταφυγίων, στη βοήθεια προς τα θύματα, προγράμματα, στις ε, γραμμές άμεσης επικοινωνίας, η προστασία των θυμάτων και των ε, και ε, νέα είδη βίας, όπως η πορνογραφία ως μέσο εκδίκησης, η παρενόχ, σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με επιφυλάξεις και αντιρρήσεις πολλών ε, συναδέλφων. Ξέρουμε πως είναι πολύ ισχυρέ από ορισμένα κράτη-μέλη και πρέπει αυτό να τα αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο. Προσβλέπω στη συνεργασία μου λοιπόν μαζί σας, στη συνέχιση μάλλον της συνεργασίας και είμαι βεβαία ότι θα βρούμε συμβιβαστικέ που θα μπορούν να υποστηριχθούν και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Okay, um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, δύο ε, για την ε, ε, παρουσίασή τους. Ξέρω ότι προχωράμε σε μια διαδικασία λογική όσον αφορά τις τροπολογίες. Να ευχαριστήσω πάντως τις εισηγήτριες. Ο κύριος Άλμπρεχτ θα μιλήσει εξ ονόματος των Πρασίνων. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων και εξ των δύο αντιστοίχων ε, σκιωδών από την Επιτροπή φάμε και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, θα ήθελα να πω τα εξή. Ε, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι το πρώτο δεσμευτικό κείμενο κατά της βίας κατά των γυναικών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει οπωσδήποτε να προσυπογράψουν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, το γεγονός ότι 14 χώρες δεν έχουν καν ε, υπογράψει και η χώρα μου η Γερμανία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει την 11η ε, ε, ε, Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογραφεί η πρόσβαση μονάχα για θέματα που αφορούν το άσυλο, την δικαστική συνεργασία και για θέματα τα οποία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αφορά η υπογραφή το σύνολο ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατέψουμε τις, ε, τους ετούντες άσυλο από οποιαδήποτε μορφή ε, βίας τις ετούσες άσυλο και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε την απόφαση του Συμβουλίου. Βεβαίως η απόφαση του Συμβουλίου δημιουργεί νομική ασάφεια γι' αυτό συμφωνούμε με την εισηγήτρια να υπογραμμιστεί η νομική συμβολή της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και να ζητηθεί νομική γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ενδιάμεση έκθεση ε, για την ε, πρόσφαση στη σύμβαση. Χαιρόμαστε που έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία αυτά στη συμβαστική 8. Λυπούμεθα γιατί η οικονομική βία κυρίως δε ο συγκεκριμένος ορισμός ε, δεν ε, έχει ε, αναφερθεί στις αιτιολογικές σκέψεις. Και επίσης εμείς θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί μία από τις πηγές της βίας. η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει ε, νομοθετικό διάταγμα σχετικά με την ε, βία των, ε, κατά των γυναικών και να ξεκινήσει διαδικασίε σε παραβάση έναντι των χωρών οι οποίες δεν υλοποιούν σωστά το κείμενο αυτό. Να για να αποσαφινιστεί η νομική βάση θα πρέπει το Συμβούλιο να πάρει τις κατάλληλες θέσεις. Ε, θα πρέπει συγκεκριμένα να ενεργοποιήσει την ε, ε, ρήτρα Πασαρέλα. Χωρίς την Πασαρέλ Clause δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ρητά και στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία κίνησης εμποδίζεται για πολλά εκατομμύρια γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριο Σκρίπετ για το ECR. Σας ευχαριστώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παίρνει το λόγο για το έγγραφο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τα καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν υποστήριξη και από την αστυνομία και από το νομικό σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σας θέσω είναι το εξή. Οι γυναίκες και τα παιδιά και τα κορίτσια προστατεύονται καλύτερα με τη συνθήκη την, ε, της Κωνσταντινούπολης. Εγώ θεωρώ ότι δεν ε, προστατεύει επαρκώς η συμφωνία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο φυσικά ενδεχομένω να ενοχλεί τα κράτη σε διάφορες περιπτώσει. γιατί θα πρέπει να αλλάξουν πολλά μέτρα και να υπάρξει προστασία χωρίς ε, τη διάσταση του φύλου, να μην υπάρχει μάλλον διακρίσεις κατά των γυναικών σε ό,τι αφορά τον ορισμό και του γάμου στα διαφορά κράτη. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να τα ανθρέφουν οι γονείς τους σύμφωνα με τα ίδια και τα έθιμα των θρησκειών. Θα πρέπει να υποδεχτούμε και τους ορισμούς που προβλέπονται. Δεν είναι, πιστεύω, ότι μπορούν να εγκριθούν μηχανισμοί οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την ε, κυριαρχία των κρατών, γιατί οι τρέχοντες ε, μηχανισμοί νομίζω ότι ήδη επιτρέπουν προστασία τέτοιων ζητημάτων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις αστυνομικές δυνάμεις σε κάθε κράτος μέλος, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση των ε, ατόμων στον ζητικό κλάδο. Αυτά όλα δεν κατοχυρώνονται στη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και τονίζω ότι δεν δεσμεύονται τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη συνθήκη αυτή και ειδικά σε ό,τι αφορά την κύρωση. Αναρωτιέμαι, η Τουρκία που έχει επικυρώσει έχει λιγότερη βία κατά των γυναικών. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει καμία επιρροή στα ποσοστά βίας οι βουλευτές επίσης ε, φαίνεται, η πολιτική φαίνεται ότι είναι κατά Υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση